Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να εξεκινήσουμε τώρα με την ημερήσια διάταξη. Τέταρτο σημείο. Έγκριση πρακτικών. Της 23ης-24ης Μαρτίου. Σχόλια. Εγκρίθηκε. Σημείο 5. Πιθανή επέκταση δείξεων προελεύσεως και της προστασίας αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μη γεωργικά προϊόντα με την κυρία Ροζιέρ. Σας ευχαριστώ. Σας παρουσιάζω λοιπόν σήμερα το προσχέδιο έκθεσης προς την Επιτροπή μας, το οποίο λαμβάνει υπόψη και αναδεικνύει μάλλον ότι πολλά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντλούν την αξία τους από την ε, προελευσή τους, από την τεχνογνωσία που υπάρχει στη χώρα προελευσή τους. Αρωτικά προϊόντα, ε, προϊόντα κλωστή και άλλα. και τα οποία αντικατοπτρίζουν και τις πολιτιστικές παραδόσεις και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γι' αυτόν τον λόγο τα αναζητούν και τα επιλέγουν οι καταναλωτές. Δυστυχώς όμως πολύ συχνά αυτή η ταυτότητά τους ε, την ε, σφετερίζονται άλλοι παραγωγή. Και αυτό δημιουργεί δύο προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, οι καταναλωτέ δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα υψηλή ποιότητα ε, προϊόντα. Και δεύτερον, οι επιχείρησει που παράγουν αυτά τα υψηλή ποιότητα προϊόντα ε, υφίστανται μια ζημιά στην εικόνα τους από τα προϊόντα μαϊμού που κυκλοφορούν με το ίδιο όνομα. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, θεωρήσει ότι είναι απαραίτητο εδώ και πολλά χρόνια, μια από το 1992 συγκεκριμένα, ε, να αναφέρεται η γεωγραφική προέλευση των τροφίμων. Ωστόσο, για άλλα προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα δεν υπάρχει καμία, κανένας είδους προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τίθεται λοιπόν το ζήτημα σήμερα, μήπως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σχέδιο. Τα μισά κράτη-μέλη, 15, έχουν νομική προστασία, παρέχουν νομική προστασία για την ε, γεωγραφική προέλευση μη ε, με προϊόντων που δεν είναι τρόφιμα. Το 2013 δημοσιεύτηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια έκθεση που έδειχνε την κατάσταση ως έχει και εξέτασε κατά πόσο θα ήταν σκόπο να δημιουργηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα. Το συμπέρασμα ήταν ότι το σύστημα που έχει δημιουργηθεί από τα μισά κράτη-μέλη αυτά τα 15 δεν είναι ικανοποιητικό. Γιατί τα μέτρα προστασίας είναι πολύ διαφορετικά. Ορισμένα ε, είναι, βασίζονται στα εμπορικά σήματα, αλλά στην ατυχητοθεσία. Διαφέρουν λοιπόν από ε, χώρα σε χώρα. Α, κάποιες, κάποια κράτη-μέλη έχουν επιλέξει, για παράδειγμα, να προστατεύουν συγκεκριμένους κλάδους, άδες, συγκεκριμένες περιοχές. Και το σύστημα συνολικά, εάν το δούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι υπερβολικά περίπλοκο. Ενώ αντιθέτω, εμεί θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα απλό σύστημα γιατί οι επιχειρήσει που παράγουν τέτοιου είδου προϊόντα, κατά τη μεγάλη του πλειονότητα, είναι μικρομεσαίε και αντιμετωπίζουν από αυτήν τον κατακαιρματισμό της νομοθεσίας ε, προβλήματα υψηλού και ανταγωνισμό. Η οθέτηση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενός κοινού συστήματος θα μπορούσε να ενισχύσει τους παραγωγούς τέτοιων προϊόντων με τοπικές ιδιωτερότητες και θα βοηθήσει τους παραγωγούς στις διάφορες περιοχές που έχουν αυτές τις, αυτά τα ειδικά προϊόντα και θα τους δώσει τη δυνατότητα να τα διαφημίσουν καλύτερα, θα τους ε, ενισχύσει οικονομικά. Και αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία να αναλογιστούμε ότι αυτές οι περιοχές συνήθως είναι ε, περιοχές αγροτικές, της περιφέρειας, με δυσκολίες οικονομικές κατά τα άλλα. Ένα άλλο θετικό στοιχείο θα ήταν η ενίσχυση του τουρισμού προς αυτές τις περιοχές. Χρειάζεται λοιπόν ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για την αναγνώριση αυτών των προϊόντων στο ευρωπαϊκό επίπεδο και θα βοηθήσει επίσης και τις εξαγωγές. Στη Γαλλία το 25 Μάλλον έχει υπολογιστεί ότι η αύξηση των εξαγωγών προϊόντων κλωστοϊφαντουργία θα μπορούσε να φτάσει το 25% εάν υπήρχε αυτή η προστασία της γεωγραφικής προέλευσης. Ταυτόχρονα οι πολίτες, οι καταναλωτές μας ζητούν καλύτερη χνηλασιμότητα, θέλουν να γνωρίζουν από πού προέρχονται τα προϊόντα που αγοράζουν, πώς έχουν ε, μεταποιηθεί, πώς έχουν κατασκευαστεί και από πού ήρθαν οι πρώτες ύλες. Η έκθεση λοιπόν της Επιτροπής ανέδειξε το πρόβλημα ότι το ο κατακαιρματισμός και τα πολλά διαφορετικά συστήματα νομικής προστασίας δεν είναι αποτελεσματικό. Γι' αυτό χρειάζεται να αναλυφθεί δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο. Το κοινό πλαίσιο αυτό θα έπρεπε να είχε τα εξή κύρια χαρακτηριστικά. Δεν πρέπει να κάνουμε απλώς μια σύνθεση, μια, μια να τα συλλογή των επιμέρους εθνικών συστημάτων. Αντιθέτως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα με κοινή, ε, κοινές αρχές και διατάξεις. Πρέπει επίσης να προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε υπερβολικά μεγάλη γραφειοκρατία και διοικητικό άχθος, γιατί όπως σας είπα απευθυνόμαστε κυρίως, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης το σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει την διαφάνεια και να μην εισάγει δημιουργεί διακρίσει μεταξύ των επιχειρήσεων. Οποιαδήποτε επιχείρηση πληρεί τι προϋποθέσεις θα πρέπει να μπορεί να κατοχυρώσει το προϊόν τη. Και τέλος να χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα ω μοχλός ανάπτυξη για τις ε, περιφέρειες της ε, Ένωσης. Τέλος, υπάρχει και το ζήτημα τη πνευματική ιδιοκτησία. ή επίσης της προστασίας ε, ε, ε, εμπορικών σημάτων. Θα πρέπει να φροντίσουμε το οποιοδήποτε νέο σύστημα υιοθετηθεί να μην αντικρούει αυτά τα υφιστάμενα συστήματα προστασίας και να συνεπάρχει ερμονικά με αυτά όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης. Έχει επίσης υπολογιστεί ότι θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 2,8% η απασχόληση στις περιοχές αυτές εάν υπάρξει προστασία των προϊόντων. Μετά από 10 χρόνια εφαρμογής ένας παρόμοιου συστήματος ε, σε συγκεκριμένη περιοχή φάνηκε ότι δημιουργήθηκαν χίλιε θέσει εργασία και αναμένουμε ότι κάτι παρόμοιο θα γίνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, θα θέλω να σα ζητήσω να υποστηρίξουμε αυτό το την πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, μια, ένα σύστημα αναγνώρισης αυτής της ε, ιδιαίτερης τεχνογνωσίας και της ιδιαίτερης ε, ιδιαιτεροτήτων των τοπικών προϊόντων. Μέχρι 28 Μαΐου μπορούν να υποβληθούν τροπολογίες. Μετά τους επόμενους μήνες θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και ελπίζω αμέσως μετά το, τη διακοπή για το καλοκαίρι, τις καλοκαιρινές διακοπές, να έχουμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και θα περάσουμε στους σκιώδεις ηγητές ή τους αντικαταστατές τους. Ο κύριος Λουίς Δεγκράντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο σκιώδης ηγητής του ΕΛΚ είναι απόν, ζητά συγγνώμη και μου ζητάει να τον αντικαταστήσω. Επομένως τα λόγια που θα ακούσετε κυρία εισηγήτρια δεν είναι δικά μου λόγια, είναι του σκιώδους εισηγητή. Ε, χαίρομαι πάντως πάρα πολύ που θα τα εκφράσω εγώ, γιατί συμμερίζομαι απόλυτα τα όσα μου, μου λέει. Συμφωνώ με τα κριτήρια τα οποία ενέπνευσαν αυτή την έκθεση. Η έκθεσή σας είναι πολύ λογική, έτσι μου είπε. Και βεβαίως μπορεί να υπάρξουν τροπολογίες που μπορεί να βελτιώσουν την έκθεσή σας, αλλά έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία ε, και αξίζει να την υποστηρίξουμε. Τα γεωργικά προϊόντα μας απασχολούν εδώ, σε αυτή την αίθουσα τα θέματα των εγγυήσεων, τη ταυτότητάς τους, τα θέματα ανταγωνισμού, ε, πώ θα τα καταστήσουμε πιο ελκυστικά. Όλα αυτά είναι στοιχεία και είναι τμήμα της ε, πλούσιας παράδοσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η οποία δεν έχει εναρμόνιση. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα ανάλογα με τη χώρα ή την περιφέρεια η οποία θέλει να υπερασπιστεί τι ιδιαιτεροτητε του Μια εναρμόνιση, αναμφίβολα, σε αυτή την περίπτωση, κατά την άποψη του ε, σκιώδου συζητητή, ε, θετική. Και εγώ συμφωνώ, θα ήταν θετικό. Αυτό γιατί, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται πολύ λογικά αυτού του τύπου τα προϊόντα ε, και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, θέμα το οποίο δεν είναι ίσονος σημασία, αντίθετα πολύ σημαντικό. Για αυτά τα προϊόντα λόγω του πλούτου τους είναι αυτά που στηρίζουν τον τουρισμό και την οικονομία, ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Επίσης θα ήταν πολύ καλό κάτι τέτοιο για τον καταναλωτή, γιατί θα είχε ένα σημείο αναφοράς, ε, εμπορικά σήματα τα οποία θα του δίναν εγγύηση. Και δεν θα έπαιρνε... Δεν θα παίρναγαν, ας πούμε, προϊόντα της πλάκας, ε, δεν θα περνόντουσαν για καλά προϊόντα, όπως λέμε έτσι, λαϊκά, για να το πω. Όλα αυτά λοιπόν θα ήταν εγγύηση ποιότητας ε, για τον καταναλωτή. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που κάνετε εσείς ε, και που μας βρίσκει σύμφωνους. Θα πρέπει αυτό να είναι συμβατό με τις παλιότερες ενδείξεις που υπάρχουν σε περιφερειακό επίπεδο και που είναι ε, τα σήματα αναφοράς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αλλιώς θα καταστρέφαμε με την εναρμόνιση αξίας, πολιτιστικές, κοινωνικές κτλ. που έχουν υψηλότατη αξία και είναι σημεία αναφοράς. Επομένως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ε, σήματα και αναφορές ε, με την ε, εναρμόνιση καταστρέφοντας τα παλιότερα, τις παλιότερες αξίες. Ό,τι αποτελεί στοιχείο ας και αναγνώρισης των προϊόντων. Επομένως, θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Συγήτρια. Θα σας υποβάλουμε ενδεχομένως κάποιες ε, τροπολογίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την έκθεσή σας. Πάντως, η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή, κατά την άποψη του Σκεωσίτη και τη δική μου. Σα ευχαριστώ κύριε Δεγκράντε. Κύριο Σαμπάτσικη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τη θα μιλήσω στη μητρική μου. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Οζιέ για την έκθεσή σας, της, για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και τις ευρωπαϊκές αξίες. Βλέποντας τις διάφορες εθνικές νομοθεσίες που αναφέρονται σε μη γεωργικά προϊόντα, φαίνεται ότι υπάρχει κενό. Ότι δεν έχουμε την νομοθεσία που θα μας επιτρέψει να προστατεύσουμε αυτά τα ιδιαιτερότητες και αυτές τις αξίες. Θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να έχουμε περισσότερες πρότυπα ευρωπαϊκά, τα οποία θα μας επιτρέψουν να εναρμονίσουμε την εθνική μας νομοθεσία μεταξύ των κρατομελών και αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο το να προσπαθήσει κάποιος να επιβάλλει ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Σε ορισμένες ε, χώρες η... εγγραφή εμπορικού σήματος μπορεί να κοστίζει ακριβά ή μπορεί να μην υπάρχει μητρό Γι' αυτό θα ήθελα να σε συγχαρώ για το γεγονό ότι προτείνεται να δημιουργηθεί ένα, μια υποχρεωτική ε, καταγραφή των εμπορικών, των διακριτικών σημάτων που χρησιμοποιούν αυτά, τα προϊόντα. Πάντως πιστεύω ότι και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα φυστάμενα συστήματα όπου υπάρχουν. Επίσης, πρέπει να δούμε τι θα γίνει όταν υπάρχει σύγκρουση και δύο διαφορετικά προϊόντα χρησιμοποιούν το ίδιο διακριτικό τίτλο, το ίδιο όνομα. Τι θα κάνουμε τότε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Président. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μελέτησα το κείμενο με πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι οι γεωγραφικές ε, ενδείξεις έχουν προσφέρει πολλά στην προστασία των ε, γεωργικών προϊόντων. Άρα θα πρέπει να αναζητήσουμε και τέτοιες προσεγγίσεις για μη γεωργικά προϊόντα. Ε, παραδείγματι στη Γαλλία έχουμε τη σταπισερή του και άλλα που είναι πάρα πολύ γνώστα σε όλο τον κόσμο. Είναι σημαντικές, ε, σημαντικά τα επιχειρήματα, η καταπολέμηση καταρχάς της παραποίησης, η καλύτερη ενημέρωση για τον καταναλωτή, ο οποίος τώρα διεκδικεί καλύτερη γνώση της προέλευσης του προϊόντος και ζητάει τοπικά προϊόντα είναι κάτι το οποίο πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη αλλά και οικονομικό συμφέρον γιατί αναμφίβολα εάν μπορέσουμε να θεσπίσουμε αυτές τις γεωγραφικές ενδείξεις θα βελτιωθεί σημαντικά όχι εξεργασιών πολλών από τις επιχειρήσεις μας θα βελτιωθεί και η εμπορική τους εικόνα ο καταναλωτικός, ε, η καταναλωτική προτίμηση κτλ. Φυσικά τίποτε δεν είναι τέλειο. Και σε αυτό θα ήθελα να πω ότι εν προκειμένου πρέπει να κοιτάξουμε τον ευρύ ορισμό της γεωγραφικής ένδειξης που μας προτείνει το κείμενο, γιατί το εδάφιο που αφορά το πεδίο εφαρμογή είναι ασαφές και ίσως με τις τροπολογίες θα ήταν σκόπιμο να διευκρινιστεί περισσότερο σε τι πρέπει να είναι διασταλτική αυτή η εφαρμογή για να χρησιμοποιήσω τη λέξη που χρησιμοποιεί το κείμενο. Και επίση πρέπει να κοιτάξουμε και την εθνική νομοθεσία όπου ισχύει. Μερικέ φορέ το καλύτερο είναι εχθρό του καλού. Δεν πρέπει δηλαδή επιδιώκοντα προστασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να ανατρέψουμε προστασία εθνική εμβέλεια, η οποία όμω έχει αποδειχθεί μερικέ φορέ αποτελεσματική. Σε αυτό θα επιμείνω, κατά τα άλλα το κείμενο το κρίνω θετικά. Κύριος Φως, ευχαριστώ. Κύριος Άντερσον. Eh, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια η οποία προτείνει την επέκταση των ε, γεωγραφικών ενδείξεων σε μη γεωργικά προϊόντα. Παρακολουθώ λοιπόν, ενημερώνομαι και διαρωτώ με πάνω απ' όλα ποιος αντλεί πλεονέκτημα και τι πιθανά ωφέλη μπορούμε να έχουμε ως προς το κόστος όμως του συστήματος. Πρέπει το σύστημα να είναι θετικό για όλους. Πρόεδρος Κοιτάξτε, έχουμε ένα μικρό θέμα ως προς την ε, διερμηνία. Κάτι δεν είχαμε προβλέψει μάλλον, ε, δεν προβλεπόταν μάλλον, ε, ίσως θα ήταν καλύτερο να προσπαθήσετε να τα ξαναπείτε. Καλώς, ε, τότε θα προσπαθήσω στα αγγλικά, μια και δεν προβλεπόταν ε, διερμηνία από τα σουηδικά. Θα προσπαθήσω λοιπόν και πάλι να ευχαριστήσω την εισηγητρία γιατί ο έργο της ε, δεν θεωρώ πως ήταν καλή ιδέα απαραίτητα. Δεν είμαι πεπισμένος ότι είναι απαραίτητα καλή ιδέα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν ποιος κερδίζει από την επέκταση στα μη γεωργικά προϊόντα των γεωγραφικών ενδείξεων και βεβαίως πόσο θα κοστίσει η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. Μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα επαφελές στο όλον του, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο διάβολος κρύβεται, ο σατανάς κρύβεται στις λεπτομέρειες. Θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσει το σημείο 18 λεπτομερέστερα η συγγετρία. Εκεί δηλαδή όπου προτείνει τη δημιουργία μιας κατηγορίας γεωγραφικών ενδείξεων εφάπαξ, με εφάπαξ τέλος. Αυτό είναι ένα σύστημα που γνωρίζουμε από τα γεωργικά προϊόντα. Όμως τα γεωργικά προϊόντα δεν είναι το ίδιο με τα μη γεωργικά. Και δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι δεδομένο πως δεν θα χρειάζεται τέλος ανανέωσης ε, στη λειτουργία αυτού του συστήματος για τα μη γεωργικά προϊόντα. Για το σήμα, παραδείγματι, το εμπορικό σήμα υπάρχει τέλος επαναληπτικό, γιατί να μην υπάρχει και για τα μη γεωργικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άντερσον και στο συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, που δεν προβλεπόταν η γλώσσα σας. Τα καταφέρατε όμως μια χαρά και σε άλλη γλώσσα. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια για την προσπάθειά της και να απαντήσω ταυτόχρονα στον κύριο Άντερσον για το ποιος μπορεί να κερδίσει από την έκθεση. Κερδισμένος θα βγει ο καταναλωτής κύριε συνάδελφε, αλλά και ο παραγωγός. Διότι ο παραγωγός χρειάζεται να έχει προστασία για το προϊόν του. Ας κοιτάξουμε και την έκθεση που μας έχει προτείνει η Επιτροπή. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το 97% των καταναλωτών ζητούν να γνωρίζουν από ε, ποια είναι τα προϊόντα που καταναλώνουν και όχι μόνο τα τρόφιμα. Και έχει δικαίωμα καταναλωτής να γνωρίζει τι καταναλώνει. Ε, ρούχο είναι, αυτοκίνητο είναι, οποιοδήποτε άλλο καταναλωτικό αγαθό είναι, θέλει να ξέρει από πού προέρχεται. Γι' αυτό θέλουμε ενιαία ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη γεωγραφική ένδειξη. Γιατί αυτό που σημαίνει σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζει μια εικόνα πάρα πολύ διαφορετική. Υπάρχουν χώρες που είναι πολύ αυστηρή η νομοθεσία. Στη Ρουμανία Φερρυπίν. Αλλά χρειάζεται να κοιτάξουμε πιο συγκεκριμένα όλη την εικόνα και να γνωρίσουμε καλά τι καταναλώνουμε. Βεβαίως και δεν θέλουμε τις ε, ε, την επιβάρυνση, τη γραφειοκρατική και όλα αυτά, αλλά πρέπει να ξεδέψουμε και τα, και τα προϊόντα μας, τα βιομηχανικά ή βιοτεχνικά. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάτι να μας πει, παρακαλώ. Πού είσαστε? Yes, thank you, Chair, and um, thanks. Uh, ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα με και εμείς από την πλευρά να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για αυτό το προσχέδιο έκθεσης και να καλωσορίσουμε και όλες τις παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών που ακούσαμε. Πράγματι το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και η Επιτροπή επιθυμεί να το αντιμετωπίσει. Και σε αυτή την προσπάθεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς επίσης και άλλα θεσμικά όργανα όπως η ΟΚΕ και η Επιτροπή των Περιφερειών, μπορούν με τη συνεισφορά τους να μας βοηθήσουν. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιος είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει να αφουγκραστούμε τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, να καταλάβουμε τις διάφορες παραμέτρους του ζητήματος, πώς θα δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο δεν θα αυξάνει δυσανάλογο το διαχειριστικό άχθος, πώς θα μπορεί να συνεπάρχει ερμονικά με τα εφιστάμενα συστήματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα συστήματα ε, καταγραφής διακριτικών σημάτων. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι όλοι πρέπει να συνεργαστούμε σε αυτή την ε, προσπάθεια, σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Η συγκεκριά παρακαλώ. Θα είμαι σύντομη κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις που μας έκαναν που έκαναν και την υποστήριξη που εξέφρασαν. Τώρα να απαντήσω σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Ναι, ε, έχετε δίκιο ότι είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε την συνύπαρξη και με τα εμπορικά σήματα, καθώς επίσης και με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με εθνικά συστήματα γεωγραφικής προέλευσης όπου υπάρχουν. Νομίζω ότι αυτό θα είναι και το πιο δύσκολο σημείο και το πιο ενδιαφέρον σημείο της όλης της Τώρα όσον αφορά την, την, ε, το κατά πόσο είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί αυτό το σύστημα, αυτή τη στιγμή το ζητούν οι επιχειρήσεις, το ζητούν και οι καταναλωτές. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι ε, υπάρχει αυτή, αυτό το αίτημα, το στο ερώτημα ποιος θα κερδίσει και ποιος θα ζημιωθεί, ε, λέω ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα με το οποίο κανείς δεν θα ζημιωθεί αλλά αντιθέτως οι επιχειρήσεις οι οποίες θα επιλέξουν να ακολουθήσουν αυτό το σύστημα περισσότερη διαφάνεια και αναγνώριση της ποιότητας των προϊόντων τους θα κερδίσουν σε καταναλωτική πίστη για παράδειγμα. Όσον αφορά για το επαναληπτικό τέλο, και το κατά πόσο θα χρειάζεται να πληρώνει μια επιχείρηση χρήματα για να ανανεώσει αυτό το διακριτικό τίτλο, Εδώ δεν μιλούμε για κάποιο είδου ιδιοκτησία υπό την έννοια τη πνευματική ιδιοκτησία ή κάτι άλλο. Μιλάμε περισσότερο για ένα είδο ε, σήμανση ποιότητα. Και το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο ε, σύστημα ελέγχου ποιότητας θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια διαδικασία για να ανανεώνεται ή να ελέγχεται κατά δηλαδή πόσο αυτό το σύστημα ελέγχου ποιότητα συνεχίζει να ισχύει και συνεχίζει να το ακολουθεί η επιχείρηση, αλλά με αυτή τη φιλοσοφία. Όχι με τη φιλοσοφία τη ανανέωση ε, ε, του δικαιώματο σε κάποιο είδου πνευματική ιδιοκτησία που θα μα οδηγούσε στη φιλοσοφία των επαναληπτικών δικαιωμάτων. Ε, τελών. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ του συναδέλφου, ευχαριστώ και την Επιτροπή για τι παρατηρήσει και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Κατάθεση τροπολογιών έως τις 28 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, για να είμαστε σαφείς. Και κλείνω το θέμα αυτό για να περάσω στο επόμενο της σημερινής διάταξης, το οποίο είναι κάπως ασύνηθες. Έχει τον αριθμό 18. Εξέταση μιας, ενός σχεδίου εκθέσεως, ετήσεις εκθέσεις του 2012-2013 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα με εισηγητή τον κύριο Σάιατ Κάριν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τώρα το σημείο της ημέρας της διάταξης γιατί αυτό με διευκολύνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ο καιρός να εξετάσουμε την τέταρτη ε, έκθεση σχετικά με τον αρχή της επικουρικότητας και αναλογικότητας που έχω προετοιμάσει και έχω τη χαρά να παρουσιάσω στους συναδέλφους. Προσπάθησα να απαντήσω να ασχοληθώ με μια σειρά ζητήματα. Πρώτον, η επικουρικότητα και η αναλογικότητα είναι ουσιώδη στοιχεία και θεμελιώδους σημασία για την διατύπωση και την κατάρτιση οποιασδήποτε πολιτική. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εξετάζουμε ποια, ποιοι στόχοι πολιτικής μπορούν καλύτερα να επιτευχθούν σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πότε είναι ε, καλύτερα να αναλυφθεί η δράση σε ευρωπαϊκό καλυτερα να ή σε εθνικό επίπεδο ή και καθόλου. Και αυτή την εξέταση, αυτή τη συζήτηση προσπαθούμε ε, να την κάνουμε να την προωθήσουμε στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και πάρα πολύ, καλό και πάρα πολύ καιρό για να λαμβάνονται τα μέτρα στο καταλληλότερο επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει λειτουργήσει αυτό, σε ορισμένες όμως όχι και τόσο καλά. Το δεύτερο ερώτημα είναι κατά πόσον η Επιτροπή σέβεται την αρχή της επικουρικότητας και κατά πόσον, το δευτερευόντος, η έλεγχη επικουρικότητας μήπως υπονομεύουν τη δημοκρατική λειτουργία. Εγώ πιστεύω ότι οι έλεγχοι επικουρικότητας θα πρέπει να ενταχθούν όλο και περισσότερο και όσο το δυνατόν πιο νωρί στην διαδικασία την ομοθετική. Γιατί ένα από τα σημαντικότερα αιτήματα, οι διαμαρτυρίες που διατυπώνουν τα εθνικά κοινοβούλια είναι ότι δεν έχουν λόγο στην αρχή της κατάρτισης της νομοθεσίας. Από την αρχή έχουν την αίσθηση ότι τους φέρνουμε πρωτετελεσμένων γεγονότων και δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους αρκετά ε, έγκαιρα. Και νομίζω λοιπόν αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη όχι μόνο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά επίση και η εμπιστοσύνη των πολιτών προ την Ευρώπη. Και είναι επίση και ζήτημα και ποιότητα τη νομοθεσία. Επίση. Διαπιστώνω ότι οι αξιολογήσει αντικτύπου που δια... Ε, ε, ε, προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το ζήτημα τη επιθωρικότητας και αυτό είναι ένα από τα θέματα που έθιξε και το Συμβούλιο ε, για τις αξιολογήσεις αντικτύπου. Επομένως αυτό πρέπει να βελτιωθεί. Έχει γίνει κάποια πρόοδος, αλλά πρέπει να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο κατατίζει αυτές τις αξιολογήσεις αντικτύπου η Επιτροπή. Τρίτον, το ερώτημα του ποιος είναι ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στον σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας. Είναι γνωστό ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να υποβάλουν γνώμες και να ισχυριστούν ότι έχει παραβιαστεί η αρχή της επικουρικότητας. Όμως αυτή η επίκληση της παραβίασης της επικουρικότητας είναι ένας από τους λόγους που μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη γνώμη το ε, ένα εθνικό κοινοβούλιο και αυτό ίσως δημιουργεί ε, λαθασμένη εικόνα. Διαπιστώνοντας πώς έχει λειτουργήσει ο μηχανισμός τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δηλαδή μετά την υιοθέτηση ε, της συνθήκης της Λασαβόνας και ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχουν τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια, διαπιστώνω ότι υπάρχουν ελλείψεις τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούσαν να συμμετέχουν πιο ενεργά σε διάφορε διαδικασίε, τι οποίε αναφέρω στο προσχέδιο εκθεσή μου. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν πιο συστηματικά να χρησιμοποιούν τη διαδικασία τη κόκκινη κάρτα. Θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του για να εκφράσουν τι απόψει του προ του διάφορου εισηγητέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά είναι θέματα τα οποία μα τα θέτουν τα εθνικά κοινοβούλια και μέλη των εθνικών κοινοβουλίων. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, ο υποφαινόμενος αναφερόμαστε σε ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, εννοούμε ότι αυτή η συμμετοχή τους θα πρέπει να ξεκινά όσο το δυνατόν πιο γνωρίς στην νομοθετική διαδικασία. Αλλά σε καμία περίπτωση ούτε ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συνενέσει στη δημιουργία ενό μηχανισμού αρνησικηρίας, κυρία, ενό μηχανισμού που θα έδινε στα εθνικά κοινοβούλια τη δυνατότητα να ασκούν βέτο σε ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό ε, το λέω προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Ε, εμείς αυτό που θέλουμε είναι τα εθνικά κοινοβούλια να μας εκφράζουν τις απόψεις τους όσο το δυνατόν πιο νωρίς, στην αρχή, όχι στο τέλος με ένα βέτο. Κάτι το οποίο πραγματικά θα υπονόμευε τις προσπάθειες που όλοι κάνουμε όπως, την κάνουμε, όπως τις κάνουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι αν ε, υιοθετήσουμε αυτά τα μέτρα θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη. Έχω αναδείξει στην έκθεση του 2013, είχαμε αναδείξει μάλλον το ρόλο του Ευρωπαϊκής, ε, του τρόπου μάλλον με τον οποίο συζητήθηκε το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν τα θεσμικά όργανα όταν κινήθηκε η διαδικασία της κίτρινης κάρτας. Υπάρχουν συστάσεις, ήδη το 2013, στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί αυτή η διαδικασία. Όπως είπα, πρέπει να γίνεται διαβούλευση με τα κοινοβούλια όσο το δυνατόν τεχνικά, όσο το δυνατόν πιο νωρί. Πιθανόν όταν είμαστε ακόμα στο επίπεδο της Λευκής Βίβλου που έχει εκδοθεί από την Κομισιόν. Και να χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο 2 για την αξιολόγηση της, αρχή, της αρχής της επικουρικότητας. Συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων όμω πρέπει να υπάρχει και στο τελικό στάδιο της συζήτησης της νομοθεσίας, γιατί πολύ συχνά το νομοθέτημα έχει αλλάξει κατά πολύ όταν φτάνουμε στο επίπεδο αυτό, στο σημείο αυτό. Και ε, πρέπει να υπάρχει μια δέσμευση από όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωση ότι τη θέλουμε αυτή τη διαδικασία και θα την ακολουθούμε. Θα ήθελα να συγχαρώ τη νέα Επιτροπή και τον νέο Επιτροπό κ. Τίμερμαντ γιατί το πρόγραμμα εργασιών το οποίο μας παρουσίασε αντικατοπτρίζει και ανταποκρίνεται σε αυτά που σας είπα και πιστεύω ότι θα, βελτιώσει, θα, θα φέρει βελτιώσει στη δημοκρατικότερη λειτουργία της Ένωσης. υπάρξει λοιπόν μια πρόοδο που φαίνεται στο πρόγραμμα εργασιών τη Νέα επιτροπή, αλλά τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν πολύ περισσότερο. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι ο σεβασμό τη αρχής της επικουρικότητα είναι αποτε απειλή για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το έργο που κάνουμε εδώ. αντιθετω είναι ενα τροπο να προστατευόμαστε, είναι ενα τροπο να είναι πιο αποτελεσματική η δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καμία περίπτωση όμω ένα σύστημα βέτο δεν θα βοηθούσε. εάν ακολουθήσουμε τα βήματα που περιγράφω, θα βελτιωθεί και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Ένωση και θα αντιμετωπίσουμε και το δημοκρατικό έλλειμμα, πιστεύω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την υποστήριξη που θα εκφράσετε στην εκθεσή μου και βεβαίως θα ακούσω με προσοχή τις παρατηρήσεις και τυχόν τροπολογίες που έχετε να μου προτείνετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Καρέμ. Δεν έχει τις κάνεις μέχρι τώρα το λόγο. Α, να και ένας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Καρύμ για τη θαυμάσια αυτή έκθεση. Βλέπουμε πολύ καλά ότι έχει μακρά εμπειρία και πολλές γνώσεις για τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Θαυμάσια μας τα είπε και χαίρομαι που το μέλημά του είναι πώς θα εμπλακούν περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια στην ευρωπαϊκή πολιτική. Γιατί αν θέλουμε να υπάρχει αποδοχή των ευρωπαϊκών ιδεοδών, θα πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να εμπλακούν περισσότερο και να θεωρήσουν ότι τα ευρωπαϊκά θέματα είναι και δικά τους. Χαιρετίζω λοιπόν τις προτάσεις που κάνετε για να εντάξετε σε αυτή τη διαδικασία περισσότερο τα κοινοβούλια. Μου κάνει εντύπωση το εξή γεγονό. Όταν εξετάζουμε τα θέματα επί των οποίων τα εθνικά κοινοβούλια έχουν υποβάλει γνωμοδοτήσει, δεν είναι τα ίδια θέματα. Οι ευαισθησίες είναι τόσο διαφορετικές από χώρα σε χώρα και τόσο διαφορετικά θέματα θεωρούνται θέματα επικουρικότητας που δεν μπορώ να βρω μια κλίδα ανάγνωσης ή κριτήρια για να καταλάβω, για να προσδιορίσω καλύτερα την αρχή της αναλογικότητας και επικουρικότητας. Απευθύνομαι λοιπόν στους ειδικού για να δω αν υπάρχει μια τέτοια κλίδα ανάγνωσης. Για να διευκολύνουμε τις εργασίες των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και τις δικές μας. Ευχαριστώ. Vielen Dank, Merci beaucoup, euh, Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με την κυρία Ντελβό. Για να πω στον κύριο Καρίμ, και φι, συνάδελφο και φίλο, ότι η δουλειά του είναι παραδειγματική, είναι ενδιαφέρουσα. Καταρχάς, ε, διευρύνουμε τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Διερωτώ με το εξή. Θα φτάσει μέχρι να προτείνετε για τις νομοθετικές εκθέσεις που ετοιμάζουμε εδώ στο Κοινοβούλιο να συνεργαστούμε νωρίτερα με τους ειδικού της α, αρμόδιας επιτροπής για τα θέματα αυτά στα, στις χώρες, στα κράτη-μέλη, πριν διετοιμάσουμε αυτές τις εκθέσεις, ούτως ώστε να έτσι να συναντηθούμε κάπου, να φτάσουμε ως την πηγή του θέματος. Καλό θα ήταν λοιπόν να ζητήσουμε τα εθνικά κοινοβούλια να μας υποδείξουν τους ειδικού και να μας τους στείλουν ε, στα θέματα που ετοιμάζουμε εμείς, αλλά να, μας, ε, να έχουμε αυτή την επαφή εκ των προτέρων. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι εργασίες κάνουν και τα εθνικά κοινοβούλια, και με αυτόν τον τρόπο τα εθνικά κοινοβούλια δεν θα εκπλαγούν όταν εμείς ετοιμάζουμε τα κείμενά μας ή και τους θα υποβάλουμε. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να χαλαρώσει λίγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει τάση να παραλαμβάνει κείμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που οδηγούν σε κανόνες και όχι σε πραγματικά νομοθετικά κείμενα υπό την πραγματική έννοια του όρου νομοθετικό. Κυρία Κρίστινσεν, τους επιτροπάτε. No. Thank you. Then, um... Κύριε Καρύμ, εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. μια και η Κομισιόν δεν θέλει να πει τίποτα, θεωρώ ότι όλα αυτά που μου είπε ο Φραν Τίμερ μας ισχύει. Εν τη αυτή περιπτώσει είμαι πολύ ικανοποιημένο που μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουμε άπλυτο περιθώριο να προωθήσουμε τα θέματά μας. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου, μάλλον τους δύο συναδέλφου που μίλησαν για τα θερμά τους λόγια. Τους ευχαριστώ για τι ενδιαφέρουσε ιδέε. Είναι ιδέες ε, που με βρίσκουν σύμφωνο, μπορώ να δουλέψω με αυτές. Μπορούμε να βρούμε κάποιον ορισμό για το τι είναι επικουρικότητα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να φτιάξουμε ένα πραγματικό ορισμό. Ε, και κύριε... Και ευχαριστώ και τον δεύτερο συνάδελφο για τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες. Με αυτόν τον τρόπο ε, θα μπορούσαμε να λάβουμε πραγματογνωμοσύνη, να δεχτούμε έτσι, τις απόψεις των ειδικών, τους ίδιους τους ειδικού από τα Εθνικά Κοινοβούλια και μας θα το κάνουμε αρκετά νωρίς στη διαδικασία, ούτω ώστε να φτιάξουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες θα ενσωματώνουν και τις ιδέες των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ε, στην, ε, σας ευχαριστώ και τα καλά σας λόγια βέβαια στη χώρα μου και στη γλώσσα μου όταν ε, αποδίδω σε κάποιον τον όρο ε, πεπειραζ, πεπειραμένο ε, σημαίνει ότι ε, αρχίζει να μοιάζει με ηλικιωμένο περισσότερο αλλά θεωρώ ότι στην εμπειρία μου αναφέρεται και όχι στα χρόνια μου. Μάλιστα. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν προθεσμία για την κατάσταση ανθρωπολογιών 27 Μαΐου και Στις 14 Ιουλίου πρόκειται η Επιτροπή να ψηφίσει. Στην δε Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου θα πάει. Το θέμα τουλάχιστον προς το παρόν αυτός είναι ο σχεδιασμός. Τώρα παραδίδω και πάλι στον πρόεδρό μας το μικρόφωνο για να συνεχίσει. Τα καταφέραμε πάντως από χρόνο, μια χαρά και σας ευχαριστώ για την ε, πειθαρχία σας. Uh, hello? hello, uh, Brussels. Uh, we... Καλημέρα, καλημέρα σας από τις Βρυξέλλες. Ε, αξιότιμοι μέλη της Επιτροπής, αξιότιμοι ε, επισκέπτες, περνάμε στο σημείο 7 της της διάταξης που είναι η ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Φαρίδα Σαχίτ, η ειδική συγγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την πολιτική πνευματική ιδιοκτησία και το, τα δικαιώματα στη πρόσβαση στην επιστήμη και τον πολιτισμό. Σας καλωσορίζουμε μέσω βιντεοδιάσκεψης. Ελπίζω ο δαίμονας της τεχνολογίας να μας βοηθήσει και να σας ακούσουμε καθαρά. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη ε, τιμή και ευχαρίστηση για εμένα που μου δίνετε τη δυνατότητα να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας με την ιδιότητά μου ως ειδική εισηγήτρια ε, για τα πολιτιστικά δικαιώματα του ΟΗΕ. Όχι το copyright. Θα ήθελα να σας διορθώσω κύριε Πρόεδρε. Έχω την εντολή από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να βρω ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές και ποια είναι τα πιθανά εμπόδια στην προώθηση των πολιτιστικών δικαιωμάτων και το σεβασμό τους για όλους και να παρουσιάσω τις συστάσεις μου προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συστάσεις για μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν τα κράτη μέλη του ΟΗΕ για τη βελτίωση της κατάστασης. Τώρα υπάρχουν κάποιες διακοπές στο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 um, I decided to devote my research in the year 2014-15 to the issues arising from intellectual property rights uh, in terms of the right to science and culture, by which I mean the right ο ήχος της ε, βιντεοδιάσκεψης δεν είναι επαρκής για να μπορέσει να μεταφραστεί δυστυχώς η ομιλήτρια. Life, which includes the right to access, to take part in and contribute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 That... Νομίζω ότι τα πήραμε τα μηνύματα λίγο πολύ που θέλησε να μας αποστείλει η κυρία Φαρίντα Σαχίτσα. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών και γι' αυτό θα παρακαλέσω όποιον δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει στη συνεδρίαση να εγκαταλείψει την αίθουσα. Σε ευχαριστώ θερμά.